So, take Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Εδώ έχουμε μία κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε εδώ. Και βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα θέμα ένστασης, αλλά και γενικότερα κάτι που έχει να κάνει με τις νέες κατεξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την νομοποίηση παράνομου χρήματος. Προτάθηκε η Τρινιδά, το Τομπάκο, η Σριλάνκα και την Ισία να προσθεθούν στον σχετικό κατάλογο. Χαίρομαι που έχουμε εδώ το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τζάστα κοινό Άστολα, από την Κομισιόν. Και όπως ξέρετε έχουμε εκπροσώπους εδώ των ε, τριών χωρών για την Τινησία, τον κύριο Μάμεν Ρίντα Τσαλκούν, που είναι υπουργό Οικονομικών της Τινησίας, το Στράτσι που είναι ε, ε υπουργό για τις εξωτερικές υποθέσεις στην Τινησία. Έχουμε τη Ρόντρον Πενέρα, που είναι πρέσβης της Σρι και τον Κόλιν Κόνελινγκ, που είναι πρέσβης της Δημοκρατίας της Τρινιδάδ και το Πάγκο. Ε, δεν έχουμε αρκετό χώρο εδώ στο βήμα, οπότε κάπως θα μετακινηθούμε εδώ. Πάντως, και η Επίτροπος Γιούροβα δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Έχουμε όμως δήλωση της Επιτρόπου. Και πρέπει να σας πω ότι η δήλωση αυτή δείχνει ότι σωστά εμείς θέσαμε το ζήτημα της ε, Τινησίας, της συμπερίληψης της Τινησίας στον κατάλογο δηλαδή αυτών και όχι μόνο για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε ότι δηλαδή έχουμε στενές σχέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τινησία, ότι είναι μεγάλη στρατηγική σημασία η Τινησία, ότι είναι πολύ σημαντική όσον αφορά το πρότυπο που μπορεί να προσφέρει στην περιοχή υπέρ του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά επίσης το γεγονός ότι η θησία βρίσκεται στο κατάλογο έχει να κάνει και με ένα διαδικαστικό ζήτημα επικάλυψης. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό και το λέει η δήλωση της Επιτρόπου σημειώνοντας τις τεράστιες προσπάθειες που κάνει η την όσον αφορά την νομοποίηση παράνομου χρήματος, ότι έχει δηλαδή πάρει μέτρα τα τελευταία χρόνια και μήνες, αλλά επίσης επειδή υπάρχει και ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης που καλύπτει αυτά τα θέματα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα αξιολογήσουμε. Γιατί Βέβαια και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να κάνει αυτόνομα την αξιολόγησή της. Καλό είναι λοιπόν που κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ όλοι μαζί. Και την ίδια αξιολόγηση και συζήτηση μπορούμε να κάνουμε και με τις άλλες δύο χώρες φυσικά. Πάντως εδώ βρισκόμαστε για εξαιτία της ιδιαίτερης κατάστασης όσον αφορά την Τινησία. Παρακαλώ, κύριε Μοράλης. Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο, και συγγνώμη, συνάδελφοι, που αργήσαμε να αρχίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί με το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα, διαδικαστικό. Κάποιος για διαδικαστικό ζητάει το λόγο από το βάθος της αίθουσας. Κύριε Βιέγκας, ξέρω ότι θέλετε να πείτε. Το έχουμε για την συνέχεια μετά τους συντονιστές. Οπότε, σας παρακαλώ, θα το συζητήσουμε μετά την ακρόαση που έχουμε εδώ. Θα το συζητήσουμε μετά. Θα έρθουμε σε αυτό που θέλετε να θέσετε, μην ανησυχείτε. Ναι, θα έρθουμε σε αυτό στη συνάντηση που θα έχουμε μετά από αυτή τη συνάντηση, λέει ο κύριος Μοράλες. Λοιπόν, Πρώτα θα ακούσουμε λοιπόν τη Γενική Διεύθυνση Just, κύριε Στόλα, μετά τους εκπροσώπους της Τινησίας, Σρι Λάνκα και Τρινιδά Τομπάκο. Παρακαλώ, σύντομα όλοι. Όλοι καταλαβαίνουμε τι διακυβεύεται εδώ. Η συζήτηση έχει γίνει σε διάφορα φόρα. Λοιπόν, Αστόλα πρώτα για πέντε λεπτά παρακαλώ. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξιότιμη πρόεδρε κυρίε και κύριοι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να μιλήσω για αυτή την κατεξοδότηση πράξη. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η συνεχής δέσμευση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τα δύο θεσμικά όργανα να αναγνωρίζουν την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην ε, καταπολέμηση της νομιμής στον και της ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ε, και ότι όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία της σχετικής οδηγίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες ό,τι αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας και περιμένω να συζητηθεί αργότερα το συμφωνημένο κείμενο. Η λίστα τρίτων χωρών, στο άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 9, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της οδηγίας ε, και έχετε λάβει τη δήλωση της Κομισιόν ε, για το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, η Επιτρόπος Γιούροβα σας έστειλε το σχετικό κείμενο. Θέλω να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία και ιδίω ε, αυτά που λέει ανακοίνωση για την Τινησία. Επειδή είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του σχέδιου ψηφίσματος η Τινησία. Καλώς ορίζω την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών της Τινησίας, του κ. Σαλγκούμα, όπως και το πρέσβη της Ιρλάνκα και της, ε, της, του και τον Πάγκο. Πριν από τρία χρόνια ξεκίνησαν διαβουλευσει και επισκέψεις παρακολούθηση. Στο Νοέμβριο του 2017 τα μέλη τη ε, ομάδα χρηματοοικονομικής δράση, τη ΦΑΤΦΟ κατέληξαν στο συμπέρασμα πω οι χώρε αυτέ Σρι Τεμεδά, μετά τον Πάγκο και την Ισία, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στρατηγικέ ανεπάρκειε για την καταπολέμηση τη νομοποίηση παράνομων εισόδων και χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε στι ε, σχετικέ συζητήσει στο πλαίσιο της ομάδας σχηματοοικονομικής δράσης ε, μαζί με τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αυτές οι στρατηγικές ανεπάρκειες είναι σοβαρές και αφορούν ε, κάποιους κρίσιμους τομείς. Έχουν εντοπιστεί στην Τινησία, παραδείγματο χάρη, ε, ανεπάρκειες ό,τι αφορά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, κανονισμό, μάλλον ρύθμιση και επιτήρηση χρηματοπιστωτικού τομέα, διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους, Σωστά αυτό θεωρείται και πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι μονάδες οικονομικών πληροφοριών δεν, έχουν, καλές, ε, ε, δεν έχουν ικανότητες, ε, χρηματοοικονομικές κυρώσεις για τη ε, χρηματοδότηση αποκρατίας, ΜΚΟ, ε, για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αυτές και κάποια άλλα ζητήματα. Παρόμοια τα ζητήματα στις χώρες της άλλης, Σριλάνκα, Τρινδάδη και τον Πάγκο. Για να πάρει αυτές αναγνωρίστηκαν από τις τρεις αυτές ε, χώρες, ε, οι οποίες ανέλαβαν ε, δέσμευση πολιτική σε ψηλό επίπεδο, με βάση ένα σχέδιο δράση που συμφώνησαν με την ομάδα χρηματοοικονομική δράση για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Οι χώρε αυτέ λοιπόν έχουν μπει στην κρίζα λίστα το compliance document ε, αυτής της ομάδας, όπως λέγεται, έγγραφο συμμόρφωση της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης. Μελετήσαμε τις σχετικές πληροφορίες και στις 13 ε, Δεκεμβρίου ε, οθετήσαμε τον κατεξοδότης κανονισμό για τις τρεις αυτές χώρες, οποίες προσθέτουμε στις χώρες υψηλού κινδύνου. Δυνάμει των υποχρεώσεών μας, δυνάμει του άρθρου 9 τη τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο. Σήμερα το Συμβούλιο συμφώνησε με αυτή την ε, λίστα τη Κομισιόν. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση τη Τινησίας και αναγνωρίζουμε ότι λήθησαν ε, θετικά μέτρα πρόσφατα και έτσι η χώρα μπαίνει στο σωστό δρόμο για την υλοποίηση σχεδίου δράση που συμφωνήθηκε με την ομάδα χρηματοοικονομική δράση. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει, όπω τονίζει και η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης αλλά και οι διμερείς συναντήσεις όπως στις 11 Ιανουαρίου στο Σεν Πίτερσμπεργκ ότι έχουν γίνει βήματα από την την Ισία για ένα καθεστώς στοχευμένων κυρώσεων και παρακολούθηση τη τομέα της σύνδεσης. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εντείνει την παροχή βοήθειας προς την Τινησία για την υλοποίηση των επόμενων σημείων του σχεδίου δράσης. Υπάρχει ένας κατάλογος εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν σχετικά σύντομα, άπαξ και η Τινησία επιβάλλει, υποβάλλει συγγνώμη, σχετική αίτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τινησία έχουν εταιρική σχέση προνομιακή και έχουν και ένα πλαίσιο στενή σύνδεση και συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επομένω, θα υποστηρίξει τι χώρε αυτέ ώστε Άπαξ και ε, εντοπίζονται ανεπάρκειες οι οποίες ε, όμως μετά ε, διορθώνονται, θα μπορέσει να βγάλει από την γκρίζα λίστα την Τινησία. Είμαστε επίσης δεσμευμένοι να κάνουμε μια αυτόνομη αξιολόγηση για την οποία του άρθρου 9 της 4ης οδηγίας για την νομοποίηση παρανομών εσόδων. Η Τινησία είναι μια χώρα στρατηγικής σημασίας και θα επαναξιολογηθεί το συντομότερο δυνατόν το 2018 σταματήσω εδώ γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος, αλλά με τα χάρη να δεχτώ ερωτήσεις. Ευχαριστώ, μακάρι και οι υπόλοιποι να τηρήσουν τον χρόνο τους όπως εσείς. Έρχομαι στον Μοχάμετ Σαλγκούν, τον Υπουργό Οικονομικών της Τινησίας. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, επιτρέψατε μου καταρχά να σα εκφράσω στο όνομα τη κυβέρνηση τη Τινησία τις ευχαριστίες μου στι επιτροπέ ΕΚΟΝ και ΛΥΜΠΕ και μέσω ε, ε, ημών και το Ευρωκοινοβούλιο που μα καλέσατε όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεών μα, όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματο και την ε, αντιτρομοκρατική δράση. Δύο προβλήματα κατά των οποίων αγωνίζεται η χώρα μα. Ωστόσο πρέπει να σας εκφράσω την έκπληξή μας και την ε, δυσκολία κατανόησης ε, της ε, ανακοίνωσης της Επιτροπής που αναγνωρίζει την Τινησία ως επικίνδυνη χώρα και συγκεκριμένα επί τη βάση της έκθεσης ΚΑΦΗ. Η χώρα μας είναι δεσμευμένη και προσιλωμένη σε όλες τις πτυχές καταπολέμησης όλων των προβλημάτων και δεν καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε καταχωριστεί μαζί με χώρες τις οποίες δεν χρειάζεται να αναφέρω. Ε, στο Μπαχρέιν το Δεκέμβριο, στην Αγία Πετρούπολη τον Ιανουάριο, εκφράστηκε ικανοποίηση για τις προόδους ε, της ε, χώρας μας ε, και αυτά μαρτυρούν για την προόδο μας. Η Τινησία ίδια είναι ένα από τα πρώτα θύματα της θερμοκρατίας και αντιμετωπίζουμε αυτό το δολοφονικό φαινόμενο που χτυπά τις περιοχές μας και κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με τις στρατιωτικές δυνάμεις μας αλλά και μέσω της, του μπλοκαρίσματος των περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατών. Ε, θεωρούμε πως η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θελήσει να υπερασπίζεται το, επικράτειά από αυτούς τους εγκληματίες είναι, είναι κατανοητή, αλλά είναι κοινή. Ε, είναι αδικό και αδικαιολόγητο η συμπερίληψη τη ισία σε αυτόν τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρά αυτόματα που δεν, και δεν λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της διαδικασίας ούτε τη πρόοδο που έχουμε κάνει με τον κίνδυνο να μείνουμε σε αυτό το, σε αυτό το κατάλογο ακόμα και αν τηρήσουμε τη, τα επιτεύγματά μας απέναντι στην ομάδα χρηματοοικονομική δράση. παρακαλεί ο πρόεδρο να, να, να, να μιλάτε λίγο πιο αργά θα έχετε λίγο χρόνο παραπάνω αν σας σα ζητώ συγγνώμη. Συνεχίζει ο Υπουργό Οικονομικών. Αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι ευρωπαϊκέ χώρε θέλουν να υπερασπιστούν τι επικράτειέ του από αυτού του εγκληματίε. Όμω είναι κοινή μα ε, πρόκληση και κοινό αγώνα. Γι' αυτό θεωρούμε πω είναι άδικη και αδικαιολόγητη η συμπερίληψη τη Ενησία από τον κατάλογο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και προχωράμε έναν αυτοματισμό που δεν λαμβάνει υπόψη τη δυναμική αυτή τη διαδικασία ούτε τη πρόοδου που έχουν γίνει στου τομεί αυτού. Με το κίνδυνο να παραμείνουμε σε αυτόν τον κατάλογο ε, ακόμα και αν ε, ολοκληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στην ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης. Μάλιστα, η την ε, μέσα στην επιστολή του Προέδρου της Ομάδας ε, Χρηματοοικονομικής Δράσης θεωρείται ως υπόδειγμα και η ΦΑΤΦ είναι αυτή που λαμβάνει υπόψη τις, τα βήματα της δράσης. Μάλιστα επέφερε τροποποιήσεις στο site της και η Τινησία αυτή τη στιγμή θεωρείται ως δικαιοδοσία υπό εποπτεία. Και γι' αυτό η ΦΑΤ δεν ζητά ε, αυξημένα μέτρα επαγρύπνησης. Τεχνικές διευκρινήσεις για το καθεστώς της χώρας μας λοιπόν και ε, που θεωρείται ένα στεναρό, ένα ισχυρό μήνυμα όπου η εύνοιά σας θα εκτιμηθεί. Ε, η χώρα μας, η κυβέρνησή μας ε, είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε. Σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε για συγκεκριμένο και λεπτομερές ορνοδιάγραμμα και συνεχίζει να το εκτελεί για να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης μέχρι, μέχρι μάλλον το αργότερο τον Απρίλιο του 2018. Τα μέτρα αυτά έχουν εκτεθεί στην ομάδα δράσης στη διάρκεια της συνόδου στην Αγία Πετρούπολη και μάλιστα μέσω μιας ε, ε, ε, απόφασης όπου λαμβάνονται οικονομικές κυρώσεις κατά των τρομακρατών. Το σύστημα ε, πληροφοριών μας ε, ε, συμμετέχει πλήρως. Χαρτογράφηση δε των κινδύνων, των οικονομικών κινδύνων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Η προετοιμασία της Επιτροπής Προσανατολισμού του ομάδας πληροφοριών όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές έχει ξεκινήσει. Η Τινησία επίσης θα δώσει μέχρι το τέλος του Απριλίου τις απαραίτητες τροπολογίες όσον αφορά το ε, Μητρό Επιχειρήσεων και επίσης όσον αφορά τα μέτρα για τη μην εξάπλωση των, των ε, όπλων μαζικής καταστροφής. Έχουμε πετύχει την αναβάθμιση δε της βαθμολογίας μας στην τελευταία σύνοδο του ΦΑΤΦΑ στο Μπαχρέιν. Η σχετική έκθεση δημοσιεύθηκε στις 6 Δεκεμβρίου, δηλαδή μία εβδομάδα πριν από τον προβλεπόμενη ε, ημερομηνία. Θεωρούμε πως έχουμε ήδη διορθώσει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις. Η Τινησία είναι σύμμορφη στις 26 από τις 40 συστάσεις της ε, ΦΑΤΦΑ και μάλιστα όσον αφορά το πάγαμα των ε, περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατών ε, ακολουθούμε τις συστάσεις και είμαστε και επίσης σύμφωνοι με τις διατάξεις του άρθρου 9 της 4ης σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Οι εμπειρογνώμονες της ΦΑΤ έχουν ήδη διαπιστώσει ότι υπάρχουν απτές προόδοι από το 2016 και ποιόν σας επαναλαμβάνω τη δέσμευσή μας να ολοκληρώσουμε όλες τις συστάσεις της ΦΑΤ μέχρι τον Απρίλιο του 2018. Η Κομισιόν ενώ δέχεται ότι δεν έχει εκτιμήσεις από τις τρίτες χώρες μέσα σε αυτή τη μεθοδολογία και προβλέπει απέναντι στην Τινησία μέτρα αυξημένης επαγρύπνησης και έτσι βλάπτει όχι μόνο τις έντονες οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις χώρε σας και τη δική μας, το, σχεδόν 80% των συναλλαγών γίνονται μεταξύ των χωρών μας, αλλά και την ε, πλήτη, τη διαδικασία μετάβασης, μεταρρύθμισης που είναι λίγο ε, ακόμα εύθραυστη. Η Τινησία έχει δεσμευτεί στη στρατηγική της σχέση με ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ξεκινήσει μια διαπραγματεύσεις για μια εις βάθος ε, εταιρική ε, σχέση χωρίς διαμεσολαβητή ώστε να δοθεί νέα όθηση. Γίνεται μια στιγμή που η στρατηγική σχέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τινησία καθιστά την τη χώρα μας την πρώτη χώρα όπου έχουμε συμφωνία ε, σύνδεσης με στόχο να βρούμε την λύση ε, των προβλημάτων Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας είναι η ολοκλήρωση πριν το πέρας του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ε, την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας είμαστε πεπισμένοι ότι οι ελλείψεις ε, της νομοθεσίας μας στην καταπολέμηση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και στην καταπολέμηση της δημοκρατίας θα διορθωθούν και ζητούμε από εσά που είστε οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών να αντισταθείτε, να αντιτεθείτε στη συμπερίληψη της Τινησίας σε αυτόν τον κατάλογο γιατί μπορεί έτσι να θυγεί η δημοκρατική ε, πορεία μας και ε, να πληγεί και η προνομιακή σχέση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια ιστορική σημασία στιγμή. Ευχαριστώ. Η κυρία για τη Σιλάνκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ εξότιμοι ευρωβουλευτέ η Σρι Λάγκα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στενές και εγκάρδιες σχέσεις. Πριν αρχίσετε, λέει ο πρόεδρο, έχουμε μπερδέψει λίγο εδώ τις θέσεις. Ε, δεν το κάνουμε επιτηδε που κάθεστε εκεί και μιλάτε από εκεί, απλώ δεν οργανωθήκαμε καλά εδώ στο βήμα. Δεν πειράζει, λέει ο εκπρόσωπο τη Σιλάνκα, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σιλάνκα έχουν στενέ και κάρδιε σχέσει και ανταλλαγέ ανάμεσα στη Σιλάνκα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνονται πολύ συχνά. Πριν από 10 μέρε η μεικτή μα επιτροπή συνεδρίασε στο Κολόμπο και υπάρχουν τακτικέ επισκέψει από εσά στη Σιλάνκα. Πέρυσι, Όλες οι κοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείες ε, επισκέφθηκαν εδώ τις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ε, δούνε πώς λειτουργεί η Επιτροπή σας προπολογισμών για να καταλάβουμε πώς μπορούμε πιο αποτελεσματικά κοινοβουλευτικά να οργανώσουμε τον προπολογισμό μας. Και όλα αυτά μετά από υψηλού πολιτικού επίπεδου συζητήσει ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τη Στριλόγκα, προκειμένου η τελευταία να υποφεληθεί από τεχνική αρρωγή και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμούμε όλους ιδιαίτερους λοιπόν την πρόσκληση των Επιτροπών ΕΚΟΝ και ΛΥΒΕ σήμερα στη Σιλάνκα για να έρθουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Αγαπητοί Πρόεδροι, στην ολομέλεια της ομάδας χρηματοοικονομικών δράσεων στην Αργεντινή τον Οκτώβριο του 2017 η Σρι Λεγκα ήταν από τις ε, χώρες ε, τις οποίες η δικαιοδοσία θεωρείται ότι είναι μία από εκείνες που θεωρούνται ότι ολοχεύουν κίνδυνο κλπ. Μετά την απόφαση αυτή λοιπόν της ομάδας χρηματοοικονομικών ε, δράσεων, ο πρόεδρος έστειλε δέσμευση ότι η Σρι Λάνκα θα αναλάβει όλα τα αναγκαία βήματα για να καλύψει τις αδυναμίες, την ομοθοσία της και τις ρυθμίσεις της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως προς την αντιμετώπιση της νομοποίησης παράνομου χρήματος, ε, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας κτλ. Στη συνέχεια ο δείκτης ε, διαφθοράς ε, το έδειξε ότι κάτι γίνεται ήδη έχει πετύχει τεράστια πρόοδο η Σρι στο μεταξύ. Και είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι επιτροπές σας ότι η Εθνική Επιτροπή Συντονισμού ρίστηκε από την κυβέρνηση της Σρι για να ελέγξει ακριβώς πώς προχωρούν όλα αυτά τα προγράμματα δράσης. Θέλουμε να διασφαλίσουμε και να διαβεβαιώσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι προχωρούμε προς την εφαρμογή μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί καταλάβαμε ότι επανέλαβε την ε, απόφαση της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης προκειμένου συμπεριλάβει την Σρι και τις άλλες ε, δύο χώρες στον κατάλογο αυτό αλλά η Σιλάνκα πιστεύει ότι με τους νόμους και τις ρυθμίσεις που έχει υιοθετήσει προκειμένου να αντιμετωπίσει την νομοποίηση παράνομου χρήματος και την αντιμετώπιση της νομοκρατίας θα πρέπει να επανεκτιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι απλώς να αντιγράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόφαση της FAT. Ε, πρέπει να υπάρχει η δικιά της μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να εκτιμάει σωστά και όχι να βασίζεται σε εξωτερικές πηγές και εξωτερικές εκτιμήσεις και να συμπεριλάβει με αυτόν τον τρόπο ε, χώρες στον κατάλογο αυτό. Αγαπητοί Πρόεδρε, σας διαβεβαιώ, η Σρι Λάνκα είναι έτοιμη να συνεργαστεί σε οτιδήποτε χρειάζεται προκειμένου να σας αποδείξουμε ότι η Σρι ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και τώρα περνάμε αμέσω στον πρέσβη Κόναλη που θα μας μιλήσει εκ μέρους της Τρινιδάδ και ΠΑΚΟ. Και πάλι ζητώ συγγνώμη που κάθεστε εκεί, εμείς φταίμε που δεν οργανώσαμε καλά εδώ το βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι, διατεκριμένοι ευρωβουλευτές. Είμαι εδώ για να μιλήσω σε ό,τι αφορά την κανονισμό της 13ης Δεκεμβρίου του 2017 και των 26-16-75 που συμπληρώνει την οδηγία 849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προσθήκη του Τρινιδάτ και τον Πάγκο στη λίστα των χωρών υψηλού κινδύνου για στρατηγικές ανεπάρκειες σε ό,τι αφορά το καθεστώς καταπολέμησης ε, τρομοκρατίας και αντιμετώπισης της, ε, του ξεπλήματος ε, χρήματος. Υπάρχουν απειλές λόγω της χρηματοδότησης τρομοκρατίας και του ξεπλήματος χρήματος αλλά και της χρηματοδότησης όπλων μασικής καταστροφής. Τις βλέπουμε ένα χρόνο. Είμαστε όμως δεσμευμένοι να τηρήσουμε τις συστάσεις της ΦΑΤΦ και τη μεθοδολογία της ομάδας αυτής. Έχουμε δείξει τις ε, δεσμεύσει μας με τις ε, αμοιβέ αξιολογήσεις. Έχουμε επίσης βελτιώσει με μέτρα τεχνικής συμμόρφωσης ε, τις επιδόσεις μας. Ήμασταν η πρώτη χώρα στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης Καρυφής και στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου που ολοκληρώσαμε τις αμοιβέ αξιολογήσεις. Σίγουρα πήκαμε σε αγροτογράφητα ύδατα για πρώτη φορά ετέθη το ζήτημα του κατά πόσο αποτελεσματικό το σύστημα AML-CTF. Τον Ιούνιο του 2016 ε, είχαμε την ε, δημοσίευση κάποιων, ε, από, κάποιων ερευνών. Είχαμε και τις τα πορίσματα του οδηγού, του Διεθνούς Οδηγού για το κίνδυνο ε, των χωρών, το ICRG. Είδαμε λοιπόν την πρώτη τεχνική συμμόρφωση και την εφαρμογή των μέτρων που είχαν προταθεί. Όπως σας είπα, κάναμε τη δυναμιβή αξιολόγηση στο πλαίσιο και της, ε, των πορισμάτων του ICRG. Ήταν ένας χρόνος η διάρκεια αυτής της αξιολόγησης. Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδο σε διάφορους τομείς. Εθνικό κίνδυνο, συντονισμός πολιτικής, εποπτεία, μέτρα προληπτικά και χρήση οικονομικών πληροφοριών. Η ΦΑΤΦ επίση λέει ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο πολιτική δέσμευση για την υλοποίηση των στάσεων τη ΦΑΤΦ για να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα όλες οι στρατηγικές ανεπάρκειες και να υλοποιηθεί ένα βελτιωμένο σχέδιο δράσης. Αυτό συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 16-23 Νοεμβρίου με την ICRG. Και έχουμε ορισμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη των στόχων. Πηγαίνουμε πολύ καλά σε ό,τι αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την ε, ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανεπάρκειες, θέλοντας να έχουμε επιχειρησιακούς ε, λειτουργικούς μηχανισμούς και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τροποποιήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο στοχευμένα. Έχουμε υιοθετήσει δύο σημαντικά νομοθετήματα για να αντιμετωπίσουμε τις στρατηγικές ανεπάρκειες ε, στο Κοινοβούλιο συζητούνται μάλλον αυτή τη στιγμή. Πρώτον, έχουμε ένα νόμο που τροποποιεί το νόμο μας για την τρομοκρατία και ενισχύει σημαντικά το προληπτικό μηχανισμό για να αντιμετωπιστούν ε, οι δράσεις ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να ε, θεσπιστούν μηχανισμοί για να τηρήσουμε τις εθνικές μας δεσμεύσεις. Πρόκειται για μια ενισχυμένη πλατφόρμα της προσπάθειας της χώρας μας για την καταπολέμηση της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Επίσης έχουμε ένα άλλο νόμο του 2017 που θα συζητηθεί τον Ιανουάριο του 2018 στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις παροχή αμοιβαία νομικής συνδρομής. Εδώ έχουμε σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, της πρόσβασης αυτές της πληροφορίες. Και τροποποιεί τις διαδικασίες του κεφαλαίου 11 του ποινικού κώδικα. Έτσι θα ολοκληρώνονται ταχύτερα οι δίκες και άλλες δικαστικές διαδικασίες. Υπάρχουν επίσης κάποια ακόμη πολύ σημαντικά νομοσχέδια. Είμαστε μία από τις ε, βασικές χώρες που έχουν μπει σε αυτό το έγγραφο συμμόρφωσης. Θεωρούμε όμως ότι λάθος ε, έχουμε συμπεριληφθεί ε, σε αυτό το έγγραφο, με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Το θέμα είναι να υπάρχουν πραγματικά κίνδυνοι, πραγματικοί κίνδυνοι. Και αν υπάρχουν οι χώρες θα πρέπει να καλούνται να διορθώσουν τις στρατικές ανεπάρκειες. Το έγγραφο συμμόρφωση στηρίζει, μιλάει μάλλον για τις πολιτικές δεσμεύσεις των χωρών. Υπάρχουν και τα μέτρα Enhanced Customer Due Diligence. Μπορείτε να καταλήξετε. Ναι, ένα λεπτό μου να μου δώσετε παρακαλώ, λέει ο εκπρόσωπος. Μία πρόταση σας, ε, αν μπορείτε. Γιατί πρέπει να ακούσουμε και τους συντονιστές και να απαντήσετε στα ερωτήματά Γι' αυτό μπορείτε να καταλήξετε με μία πρόταση, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ θα ακολουθήσω, θα συμμορφωθώ με τον περιορισμό που μου επιβάλλατε. Εμείς έχουμε δεσμευτεί και θα έχουμε διάλογο ε, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας σε υψηλότερο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι ζητάω το αδύνατο, αλλά παρακαλώ του συντονιστές ένα με δύο λεπτά. Όχι πάνω από δύο λεπτά ο καθένας, παρακαλώ. Για να ακούσουμε και τους συντονιστές της ΕΚΟΝ μετά. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι συντονιστές εδώ. Πέλς, πρώτα Μιλάω γερμανικά εγώ. Καταρχάς, θέλω να καλωσορίσω τους εκπροσώπους των τριών χωρών που είναι εδώ σήμερα, τον Υπουργό. Μιλάω γερμανικά εγώ. Καταρχάς, θέλω να καλωσορίσω τους εκπροσώπους των τριών χωρών που είναι εδώ σήμερα, τον Υπουργό. Ξανασυζητήσουμε για να δούμε αν θα πρέπει να αφαιρεθούν από αυτό το κατάλογο οι χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούλτς. Η κύριε Ματσόλα, δεν θέλει το λόγο. Όχι, όχι, γιατί συμφωνώ με τόσο μόλις υπόθηκαν, γι' αυτό δεν θέλω το λόγο. Ωραία. Συμφωνείτε με όλους, είπε ο κύριος Βαλτς. Καλώς. Η κυρία Σίπελ, σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Δύο λεπτά. Ε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που μπορούμε να έχουμε με τις τρεις χώρες. Για το ότι έχουν δεσμευτεί και προχωρήσει για την κάλυψη των κριτηρίων προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Όμως, δεν βλέπω προς το παρόν να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα μέτρα αυτά θα ολοκληρωθούν. Είχε μια υπόσχεση από μια χώρα μέλος που έλεγε εμεί θα είμαστε έτοιμοι τον Απρίλιο, εγώ δεν θα το εμπιστευόμουν αυτό. Ωραία, όταν θα είσαστε έτοιμοι θα το. Έχουμε καλές σχέσεις και καλή συνεργασία με τις τρεις αυτές χώρες. Με την Τινησία για παράδειγμα έχουμε προνομιούχα εταιρική σχέση. Και συνεπώς έχω κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορούμε να καταψηφίσουμε την κατεξουδότηση πράξη. Αλλά έχω και μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Έχουν και συνεπώς έχω κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορούμε να καταψηφίσουμε την κατεξουδότηση πράξη. Αλλά έχω και μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Έχουν... Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος συντονιστής, ο Ραμόν Τρεμόσα. Παρακαλώ, από την Άλντε μετά από το EDF το ECR. Ε, παίρνω το συντονιστή από κάθε επιτροπή. Δυστυχώς κάποιοι λείπουν, οπότε επόμενος ε, συντονιστής της ΕΠΟΜ, οπότε δώστε το λόγο στον κύριο εδώ. Ωραία. Επόμενος συντονιστής της Άλδη δεν θέλει το λόγο, αυτό είναι. Then I'll go to the next one. Okay, right, who's the next one then? No, let's do Tremosa and then Luke after. Right, so Tremosa first. Can you just speak? να σα πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει πια. Απλά ήθελα να παρατηρήσω ότι εν γέννη είναι πρώτα ο συντονιστής του ECR και μετά το ALDE. Αν ο κύριος Τρεμόζα θέλει να μιλήσει πριν από μένα, δεν έχω πρόβλημα. Και εγώ είμαι τη έκονα συντονιστής. Δεν θέλω να παρέμβω γιατί κάθε συντονιστή τη έκονα. Θα μιλήσετε έτσι κι αλλιώ, οπότε α λήξει αυτό το επεισόδιο. Ο Τρεμόζα είναι συντονιστή. Πρώτα ο Τρεμόζα λοιπόν και μετά τώρα που ξέρουμε. No, just uh, a very brief intervention. Λοιπόν, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στην ε, ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης. Ε, έχω μιλήσει κατάλογος αυτός προσθέτει την Τινησία, δεν βάζει άλλες χώρες που βρίσκονται στην περιοχή. Οπότε δεν το καταλαβαίνω. Έχω όμως εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτούς που δουλεύουν για την αντιμετώπιση της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Ομάδα FAT, η Γκάφη. Οπότε συμφωνώ με τον κύριο Λουκό ότι θα έπρεπε να έχουμε μία κατεξοδότηση πράξη για κάθε χώρα χωριστά. Γιατί είναι δύσκολη η σύγκριση. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γιατί ακριβώς χώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω και εγώ να κάνω μια ερώτηση, γιατί για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν με ικανοποιήσει η αρχική σας δήλωση. Βρίσκω, για να τα πω όμα, πολύ γραφειοκρατική για να αποφύγετε μία δήλωση που είναι θετική. Μιλάτε για τις αδυναμίες κτλ. τα Ωραία και λοιπόν κάποιων ζητημάτων όπως είναι το μητρό. Εγώ δεν σας ρωτάω γιατί ξέρω την απάντηση. Αν τα κριτήρια ήταν ε, ότι πρέπει να βάλετε όλες τις χώρες που δεν έχουν αυτό το μητρό, και το άλλο που λυπεί είναι ότι είναι δίκαιο απέναντι στις διαφορές χώρες. Λοιπόν, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να απορρίψουμε το αίτημά της, ας μας δώσει περισσότερα στοιχεία που να μας πείσουν. Γιατί από αυτά που είπατε στην αρχή και η δήλωση που κάνετε για να μας πείσετε, προς το παρόν δεν φτάνει. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους τρεις πρέσβες. Θα αρχίσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι. Τρία-τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Παρακαλώ. Ελπίζω να θυμάμαι τις ερωτήσεις. Αν δεν τις θυμάμαι να μου τις θυμίσετε. Πρώτα απ' όλα για το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε να πούμε ημερομηνίε ακριβώ γιατί πρέπει να ελέγξουμε την νομοθεσία. Και θα πρέπει να περάσουμε από όλη τη διαδικασία που σημαίνει να πάμε επί να δούμε τη λειτουργία κτλ. Άρα είναι και θέμα εργασίας που έχουμε να κάνουμε για, για να βγάλουμε τη χώρα από τον κατάλογο. Τώρα, όσον αφορά την αναδιγράψαμε την γκάφη ή κάνουμε τη δικιά μας αξιολόγηση. Κάνουμε την αξιολόγηση και στα τέλη της χρονιάς θα έχουμε τα αποτελέσματα που θα συμπληρώσουν τον κατάλογο της ομάδας κρηματοοικονομικής δράσης. Τώρα το θέμα του Μητρώου είναι κάτι που θα ζητά μόνο εμείς αλλά και η FAT. Τώρα γιατί την Ισία. Το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο η FAT αξιολογεί τις διάφορες χώρες συμφωνείται με τις χώρες. Και η Τινησία δέχτηκε να είναι σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Σε αυτό το ημερολόγιο λοιπόν, σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, οι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν και θα αξιολογηθούν και αυτές. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα θα δείτε και τις άλλες χώρες στον κατάλογο. Όσον αφορά την επίπτωση της ε, ένταξης αυτό το κατάλογο, δεν είναι τιμωρητική, δεν είναι για να τους εμποδίσουμε σε κάτι, δεν είναι για να εμποδίσουμε τη βοήθεια προς τη χώρα. Οπότε δεν είναι τόσο τρομερό άλλα μέτρα. και για το κατά πόσο είχαμε την πληροφορία αυτή για την αξιολόγηση, ναι, την είχαμε. Μελετήσαμε όλο το υλικό ακόμα και μέχρι σήμερα και σύμφωνα με αυτό υπάρχουν ακόμα δυναμίες και δεν πρόκειται για νούμερα. Πρόκειται για το νόημα, τη σημασία που έχουν αυτά. Ήδη απάντησα για τη Λιβύη. Είναι θέμα αργότερα. Και το χρονοδιάγραμμα για τη δικιά μας αξιολόγηση, σας είπα, θα είναι στο τέλος της χρονιάς. Τώρα τι ξέχασα. Εκτός μικροφώνου η ερώτηση. Πόσες χώρες έχουν αυτό το beneficiary register ownership στη... στον κόσμο. Εμείς με τη σειρά αξιολογούμε τις χώρες, η Επιτροπή και η FAT με το χρονοδιάγραμμα που έχει καθορίσει και εμείς αυτό κοιτάμε. Και υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχει μια ρύθμιση για την επιθεώρηση του μη χρηματοπιστωτικού τομέα και είναι και αυτή μια δυναμία που διαπιστώσαμε. Οπότε δεν είναι μόνο για το beneficial ownership, είναι και γι' αυτό. Κατά τα άλλα, σήμερα θα έχουμε ε, πράξη με διαφορετική για κάθε χώρα. Κατευθυντήριες γραμμές δηλαδή για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό δεν λέτε. Όχι, λέει η Επιτροπής. Μιλάμε για τον κανονισμό και την εποπτεία του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Ωραία. Τώρα. Λοιπόν, η πρέσβης παρακαλώ. Θα αρχίσουμε με τον Υπουργό Οικονομικών της. Ο Υπουργό τη Τινησία, η πρόοδο που έχουμε σημειώσει και συνεχίζουμε να σημειώνουμε είναι σημαντικό και θα πρέπει να το εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εξασφαλίσει έτσι ότι μένουμε στο ίδιο μονοπάτι, να έρθει σε επικοδομητικό διάλογο μαζί μα όπω και σε τόσα άλλα θέματα. Η Σρι είναι μια χώρα που έχει για την ενίσχυση της δημοκρατίας, για την ε, ε, ε, σταθεροποίηση του κράτους δικαίου. Και για αυτά τα θέματα είμαστε σε διάλογο με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και γι' αυτό θα εκτιμούσαμε, αν ληφθεί υπόψη, ότι έχει αναπτυχθεί μηχανισμός για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων για να είμαστε πλήρως σύμμορφοι με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε ξανά την ευκαιρία να πάρω το λόγο. Να πω εν συντομία ότι από τότε που έχω εγώ αναλάβει τη ως πρέσβης στην Ένωση, η σχέση μου με την Κομισιόν ήταν, είχε πάντοτε να κάνει με το πολιτικό διάλογο, τη διαβούλευση και το συντονισμό. Θα ήθελα, διαρωτώ μεθά αν αυτή η διαδικασία έχει ακολουθηθεί αυτή τη φορά. Η χώρα μου έχει έχει λάβει ε, την ενημέρωση τρεις μέρες πριν, όπου έπρεπε να απαντήσουμε. Πόσο εξ όσων γνωρίζω, το Τρινιτάρι και το Μπάκο ποτέ δεν είχε διαβούλευση με την Κομισιόν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και νομίζω, όπως και οι βουλευτές, ε, θα πρέπει να ανησυχούμε για αυτή την εξέλιξη. Δεύτερον, υπήρξε κακο, ε, κακοχαρακτηρισμός για το τι κάνουμε στη χώρα μου. Ποτέ δεν ε, σύστησε η ΦΑΤΦΟ οποιαδήποτε κύρωση σύμφωνα με τη διαδικασία του. Πώς τότε ζητούμε από αυτές τις χώρες, ε, μάλλον αυτές οι χώρες να τιμωρηθούν εφόσον το ΦΑΤΦ δεν το έχει αυτό συστήσει να γνωρίσει Τρίτον, από όσο γνωρίζω το Τριντάτι και το, και το Μπάγκο τηρεί 38 από τις 40 συστάσεις που έκανε το ΦΑΤΦ. Ε, είμαι μερικώς σύμμορφη ε, σε μεγάλο βαθμό σύμμορφοι, δηλαδή είμαστε, ε, έχουμε ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις μας παρακαλώ λοιπόν. Τρεις χώρες εδώ είναι ε, στην υπόθεση αυτή, αλλά παρακαλώ να εξετάσετε εάν έγινε διαβούλευση ή όχι και παρακαλώ να το πενεξετάσετε γιατί όπως σας είπα είμαστε σύμμορφοι με τις 38 από τις 40 συστάσεις και η ΦΑΤΦΟ ποτέ δεν σύστησε την επιβολή κυρώσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ε, μας ε, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Οι συνάδελφοι που ήρθαν για την ψηφοφορία που δεν συμμετείχαν στη συζήτηση, παρακαλώ να έχετε λίγο υπομονή γιατί θα ζητήσω τώρα από τον κύριο Γκουαλτιέρη να πει πώς θα προχωρήσουμε. Καταρχάς να ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Τινησίας, τους πρέσβεις της Σριλάνκα και του Τρινιδάτη και το Πάκο και την Κομισιόν βεβαίως. Αν και θα θέλαμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Επίτροπο Γιούροβα, αλλά εκτιμούμε ότι ήρθε η Γενική Διευθύντρια. Για να είμαι ειλικρινής, Βέβαια, τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη αξιολόγηση, αλλά ειλικρινά, εγώ δεν έχω πιστεί Ε, βλέπω να υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη δήλωση στις, δηλω... στις διάφορες δηλώσεις της Επιτροπής. Εγώ ξέρω και έχω από αυτά που ξέρω και από αυτά που ακούω, έχουμε τώρα ένα συνδυασμό έλλειψης ολοκλήρωση κάποιων στοιχείων που είναι σημαντικά αλλά που από μόνα τους δεν αρκούν για να, για να αξιολογηθεί την νησία με αυτόν τον τρόπο και εδώ έχουμε μια επικάλυψη χρονική Ανάμεσα στην πρώτη αξιολόγηση, τα μέτρα που μεταξύ έχουν ληφθεί και τώρα Έχουμε κάποιες, ε, την εφαρμογή ε, νομοθεσίας, έχουμε, έχει εκδοθεί μια κατευθύντρια γραμμή επίπεδου 2 και δύο νομοθετήματα τα οποία δεν ισχύουν σε πολλές χώρες που δεν είναι σε αυτόν τον κατάλογο. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση λοιπόν. Πιστεύω πως η Κομισιόν θα πρέπει να είναι λίγο πιο σαφής στον τρόπο αξιολόγησης και στο... να αφαιρέσει από τον κατάλογο γρήγορα με αυτόνομη κρίση. Και τι σημαίνει γρήγορα, τι θα γίνει μια μόνη ε, κατοξιδότηση πράξη. Ε, σύμφωνα με την κατάσταση αυτή θα έχουμε συμπερίληψη από την ΦΑΤΦ και από την, Κομισιό, και από την Κομισιόν. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια αξιολόγηση, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή λίγο λεφτών για να δώσουμε το χρόνο στις πολιτικές ομάδες ε, μεταξύ τους να συνεννοηθούν, να αξιολογήσουν και μετά θα αποφασίσουμε τι κάνουμε γιατί έχουμε προγραμματίσει ψήφο ψηφοφορία, η οποία πρέπει να γίνει. Ένα λεπτό, δύο λοιπόν διακοπή για να μπορέσουν οι ομάδες αναμεταξύ τους να συνεννοηθούν. Και να ζητήσω από την Επιτροπή και από τους προσκεκλημένους μας να ε, βγουν και θα ξαναρχίσουμε σε λίγα λεπτά. So, um, αυτό που εννοεί ο κ. Γουαλτιέρη είναι οι, τα, οι ευρωβουλευτές να μείνουν, οι πολιτικοί σύμβουλοι επίσης, οι κομισιόν και οι λοιποί παρακαλούμε να βγουν για λίγο. Θα λάβουμε απόφαση και θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία στη συνέχεια.